Ευχαριστώ. Ε, για τα καλά σου λόγια. Πάμε στο σημείο 6 της σημερινής ε, ημέρησης διάταξης. Κοινή συνεδρίαση με τους αντέλφους από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Αφορά την κατάσταση ασφάλειας στη Συρία μετά την ε, ανακοινωθήσα αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων. στα ε, σύνορα με το Ιράκ και την ε, Ιορδανία και τη Συρία φυσικά. Με αυτόν τον τρόπο το Ιράν δεν θα, μπορέσει, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να έχει δημιουργήσει ένα διάδρομο που θα φτάσει μέχρι το Λίβανο και να μεγαλώσει την επιρροή στην ε, επιρροή. Η Τουρκία προσπαθεί να περιορίσει την επιρροή των, ανταρτών, των Κούρδων ανταρτών και τις ε, πολιτοφυλακές τους. Και με αυτόν τον τρόπο ε, θα πρέπει να αναγκάσουμε τον Άσαντ να έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων στην ε, Γενέβη, αλλά θα πρέπει, αν το καταφέρουμε αυτό, θα πρέπει να περιορίσουμε την, τους πολεμοχαρείς στο Ιράν που θέλουν να μεγιστοποιήσουν την επιρροή. Λοιπόν, θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, ε, τι σενάρια για μετά την αποχώρηση των Αμερικανών από τη Συρία ε, και το ρόλο που θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, στη Συρία και περιφερειακά. Η κυρία Έρικα Φερέρ, τμήματάρχης της ΜΕΝΑ ε, για τη Μέση Ανατολή, Αίγυπτο, Συρία, Λίβανο και Ιορδανία και τη Λίνα Κατίμπ, θεματάρχη ε, του προγράμματος του Chatma House για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στους δύο μιλητές μας, θα ήθελα να θέσω κάποια επιπλέον ερωτήματα ε, για τη συζήτηση. Μετά από το προηγούμενο θέμα που ακούστηκε στη ΣΕΝΤΕ, ε, η Άγκυρα ε, έχει ανακοινώσει δράσεις ε, εναντίον του, της πολιτοφυλακής του YPG στη Βόρειο Συρία. η Ουάσιγκτον είπε όμως να μην προβούν σε μονομερή δράση, γιατί τις δυνάμεις αυτές στηρίζουν οι Αμερικανοί. Τώρα που αποχωρούν όμως τα Αμερικανά στρατεύματα, πώς θα μπορέσουν κάτι να αποψή σας πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί εάν παρά τις ε, προειδοποίησεις ε, η Τουρκία κάνει επιθέσεις εναντίον των Κούρδων ανταρτών. Επίσης και το ISIS παρότι έχει αποθυναμώσει στη Συρία και στο Ιράκ δεν έχει νικηθεί. Ε, και οι επιθέσεις στα αμερικανικά, βρετανικά και κουρδικά στρατεύματα το δείχνουν αυτό. Επομένω, τι θα γίνει με την αποχώρηση τώρα των Αμερικανικών στρατευμάτων από την Συρία και τι επίπτωση αυτό θα έχει στο μαχητικό δυναμικό του ISIS. Επίση, έχουμε κανένα χρονοδιάγραμμα για τα βήματα που θα ακολουθήσει η διαδικασία μετά ε, τη αποχώρηση, μάλλον. Τα βήματα τη διαδικασία αποχώρηση. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην ε, Επιτροπή. η κυρία Φερέρ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση για να μιλήσω στην, στις δύο επιτροπές. Με μεγάλη χαρά έρχομαι, ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρχομαι έρχομαστε σε επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, και είναι και εδώ η κυρία Κατήμ, η οποία γνωρίζει πραγματικά την περιοχή στη Συρία, τις προκλήσεις μετά τις πρόσφατες εξελίξεις. Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία για να δούμε πού, πού είμαστε, ποιες είναι οι προσκλήσεις και τι πολιτικές δυνατότητες, έχει, δυνατότητες πολιτικής μάλλον έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και να, θέσουμε κάποια, να δώσουμε κάποια απαντήσεις στα ερωτήματα που θέσατε. Να υπενθυμίσω ότι η βάση για την ε, ευρωπαϊκή πολιτική και τις δραστηριότητε για τη Συρία πολιτικά και σε ό,τι αφορά την υποστήριξη που δίνουμε. Θα ήθελα να σας δείξω ότι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Συρία, όπως συμφωνήθηκε τον Απρίλιο του 2017, παραμείνει ε, σταθερή, ε, ισχύει ακόμα και σήμερα και να μην ξεχνάμε τις ε, κατευθυντήριες αρχές. Χρειαζόμαστε να τελειώσει ο πόλεμος μέσω μιας πραγματικής πολιτικής μετάβασης με βάση το ψήφισμα 2254 ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Χωρίς πολιτική μετάβαση δεν θα υπάρχει βιώσιμη ασφάλεια ούτε ειρήνη. Και θα επανέλθω σε αυτό. Θέλουμε ουσιαστική μετάβαση στη Συρία με υποστήριξη της ε, πολιτικής ε, αντιπολίτευσης να ενισχύσουμε την, τις οργανώσεις των πολιτών, προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία λόγου κτλ. Βασικά ερωτήματα τα οποία θα πρέπει να απαντηθούν είναι η λογοδοσία, ε, εθνική συμφιλίωση και ε, δικαιοσύνη σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι φυσικά να σώσουμε ζωέ μέσω τη ανθρωπιστική βοήθεια. Υποστήριζουμε την ανθεκτικότητα του πληθυσμού και της κοινωνίας της Συρίας. Από αυτή τη στρατηγική απορρέουν οι πολιτικέ Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα συμπράσματα του Συμβουλίου που υιοθετήθηκαν τον Απρίλιο του, 10... του περασμένου έτου. Του 18 δηλαδή. Ποια είναι τα ουσιαστικά στοιχεία της πολιτικής αυτής και να τα εξετάσω με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις ε, και κυρίως την αναγγελία της, ε, αποχώρησης των Αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία και την, ε, το ότι οι εξτρεμιστές ε, HTS κατέλαβαν την επαρχία Γκλίμπ. Ε, και με την στήριξη των Ρώσων ε, μπήκαν οι εξτρεμιστές. Ε, μάλλον των δυνάμεων του Ασάντ. Ε, υπάρχει στην όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια, υπάρχει μια προσέγγιση σταθερή, συνεπή, ε, με βάση μια συγκεκριμένη πολιτική. πολιτική διαδικασία. Οποιαδήποτε βιώσιμη λύση στη σύγκρουση απαιτεί καταρχάς μία ειρνευτική διαδικασία που να οδηγεί σε πραγματική πολιτική μετάβαση με βάση το ψήφισμα του 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας και το ανακοινωθέν του, του, ε, του 2012 της Γενέβης θα πρέπει να υπάρχει ενότητα, ε, εθνική κυριαρχία και δαφική συνέχεια του Συριακού κράτους. Εμείς στηρίζουμε την διαδικασία του ΟΗΕ και το νέο απεσταλμένο ε, του ΟΗΕ στη Συρία. Γκέρτ ε, Πέντερσεν. Θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσει τη διαδικασία. Ο κ. Πέντερσεν ακούει, έρχεται σε επαφή με διάφορους τέρους και φορείς και θα πρέπει να δούμε αν θέλει να συνεχίσει με την ε, συνταγματική διαδικασία της Άστανα. Ε, η εντολή του βασίζεται στο ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας και πιστεύω ότι θα προσπαθήσει, θα προσπαθήσει να ξαναδεί όλα τα ευρύτερα θέματα που έχει θέσει το ψήφισμα, όχι μόνο το Σύνταγμα της Συρίας. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τη στάση του. Εμείς, στο μεταξύ, ε, δίνουμε στήριξη στην πολιτική αντιπολίτευση, την SNC, την ε, κοινωνία των πολιτών της Συρίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να παίξουν πραγματικό ρόλο στη μετάβαση, στη μεταβατική αυτή περίοδο. Είμαστε τμήμα της ε, Παγκόσμιας ε, Συμμαχίας για να καταπολεμήσουμε το ISIS και να σταθεροποιήσουμε τη Βόρεια και Ανατολική Συρία. Λοιπόν, στα βόρεια-ανατολικά της χώρας, να δούμε τι συνέπειες έχει, αλλά και στη Συρία όλο αυτό και για τους ε, εμπλεκόμενους φορείς για μια πιο λεπτομερή εικόνα ασφαλείας και τη σχέση ανάμεσα στις δυνάμεις αυτές ε, θα ακούσουμε από τους επόμενους ομιλητές. Εμείς πιστεύουμε ότι ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε θέλουν να νικηθεί το ISIS αλλά και να περιοριστεί η επιρροή του Ιράν στη Συρία που είναι βασική προτεραιότητα για κάποιους πολιτικούς εταίρους στη Ουάσιγκτον. Υπάρχουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα ακόμα σε ό,τι αφορά το ρυθμό και το πρόγραμμα για την αποχώρηση των Αμερικανών και πρέπει να δούμε ακριβώς, ε, ζητούμε διευκρινήσεις από τους ε, συμμάχους μας στην Αμερική και να συνεχίσουμε δυνατόν τις ε, δραστηριότητες σταθερότητα, ούτω ώστε να εξασφαλίσουμε στη βόρειο Ανατολική Συρία θα νικηθεί το ISIS. Ε, ίσως είναι πιο εύκολο για κάποιους από τους εταίρους να συνεχίσουν δραστηριότητες τους αυτοί όταν φύγουν οι Αμερικανοί. Ε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει κενό εξουσίας. Υπάρχουν άμεσες συνέπειες ε, μετά την αναγγελία της αποχώρησης των Αμερικανών και φαίνονται ήδη από τώρα. Η Τουρκία προς το παρόν ε, προέκυψε ως βασικός ε, αποδέκτης του ωφέλου. Ε, παρότι οι σχέσεις με του Αμερικανού ε, είναι περίπλοκες υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ Τουρκία και Ηνωμένε Πολιτείε. Να δώσουμε στην Τουρκία, ας πούμε, που δίνει μάλλον στην ε, Τουρκία την ε, δικαιολογία για να μπει στο παιχνίδι. Το STF ε, των Κούρδων, βασικά των Κούρδων, αισθάνεται απειλούμενο από την Τουρκία. οι Αμερικανοί, όπως είπατε κύριε Σέπαρτ, Ε, δεν θέλουν φυσικά οι Τούρκοι να επιτεθούν στους ε, βασικούς τους εταίρους, ε, τους Κούρδους στα βορειοανατολικά. Ε, Επίση, πρέπει να θυμίσουμε στους Τούρκους ότι πρέπει να επιτρέψουμε την πρόσβαση ανθρωπιστική βοήθεια, να προστατευτούν οι άμαχοι κτλ. κτλ. Η αναγγελία της αποχώρησης των Αμερικανών επηρεάζει επίσης την κατάσταση και την ισορροπία δυνάμεων στα βορειοδυτικά της χώρας, στο Ιντλίπ, ριζοσπαστική γύρω από το HDF, ε, βλέπουν ότι η Τουρκία εστιάζει στα βόρεια-ανατολικά και έχουν αδράξει την ευκαιρία για να διευρύνουν και να παγιώσουν τη θέση τους. Ελέγχουν πάνω από το 80% της επαρχίας του Ιντλίμπ. Ε, οι πιο μετριοπαθείς υποχωρούν με λίγη υποχώρηση, υποστήριξη από την Τουρκία και η κατάσταση είναι πολύ ασταθής. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκές επιχειρήσης ε, τις μη ανθρωπιστικές. Η αποχώρηση των Αμερικανών, η αναγγελία, ε, καθιστά τη θέση του, της Ρωσίας και του ρωσικού καθεστώτος και την, ε, των Ιρανών πιο έντονη. Ε, κινούνται οι δυνάμεις αυτές ε, στα βορειοανατολικά εν ώψη ε, της αποχώρησης των Αμερικανών και στις πετρελοπηγές Ε, βέβαια για να κατακτήσει το καθεστώς σε αυτή την περιοχή θέλει α, βοήθεια από τη Ρωσία. Η δικαιολογία θα είναι ότι θα πολεμήσουν και θέλουν να νικήσουν τους τρομοκράτες. Και τότε σε αυτή την περίπτωση υπάρχει κίνδυνος για ανθρωπιστική κρίση. Στα βορειοδυτικά διορθώνουμε. Το καθεστώς κερδίζει ε, και η Ρωσία και η Τουρκία και το Ιράν, αλλά έχουν άλλο, άλλο συγκρουόμενα συμφέροντα. Η Λίνα θα τα πει πιο αναλυτικά όλα αυτά. Θα ήθελα τώρα να περάσουμε στο γεγονός ότι το Συριακό καθεστώς προσπαθεί να ανακτήσει ε, διεθνή νομιμότητα και κονδύλια για να χτίσει τη χώρα. Ε, συμβάσεις δίνονται σε διάφορους υποστηρικτές του καθεστώτος και βλέπουμε ε, συμφέροντα, ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις. Ε, ποια είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του καθεστώτος και των συμμάχων για να ε, ανακτήσει την νομιμότητα. Είμαστε αποφασισμένοι να μην ξεχάσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί, έχει μεγάλη επιρροή σε ό,τι αφορά την αναγνώριση, ε, ομαλοποίηση και ανοικοδόμηση της χώρας. Θα ήθελα να επαναλάβω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και ξεκαθαρίζει ότι θα υποστηρίξει την ανοικοδόμηση μόνο στην περίπτωση συνολικής, πραγματικής, ε, χωρίς αποκλεισμού πολιτικής μετάβασης στα πλαίσια της διαδικασίας του ΟΗΕ και όταν ξεκινήσει πραγματικά. Δεν πρόκειται να ξεκινήσουμε σε αρχικές προσπάθειες πριν γίνουν ε, οι προσπάθειες ε, Ουσιαστικέ προσπάθειε μετάβαση υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Θα ήθελα να πω δύο λόγια για του πρόσφυγες και την επιστροφή των προσφύγων. Όπω ξέρετε, ε, ακούστηκαν εκκλήσει κυρίω από τη Ρωσία για ένα σχέδιο για την επιστροφή του. Κράτη υποδοχή ε, και η Ορδανία και ο Λίβανο, επιμένουν ότι οι πρόσφυγε πρέπει να επιστρέψουν στη Συρία. Πρέπει να ξεκαθαρίσω το εξή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει το βάρο σε αυτές τι χώρε που έχει πέσει στη Τουρκία, Λίβανο, Ιορδανία, γιατί γενναιόδωρα δέχτηκαν εκατομμύρια ε, Σύριους προσφύγους. Και δεν είμαστε κατά της ε, επιστροφής των προσφύγων, σε καμία περίπτωση. Όμως, διατηρούμε τη θέση μας, όπως ακούστηκε στα συμπεράσματα του 18, και συμφωνούμε με τα, τις αξιολογήσεις ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι πρέπει ε, να υπάρχουν οι συνθήκες ώστε να επανέλθουμε κάθε ασφάλεια, αξιοπρέπεια κτλ. και οι προσφυγές και οι εσωτερικά εκτοπιστέντες κτλ. Και, και αυτό δεν υπάρχει ακόμα. Γιατί υπάρχουν δολοφονίες ακόμα κτλ. Ε, προβλήματα ασφάλειας τα λοιπά και δεν είναι όριμες συνθήκες. Ε, το καθεστώς και η Ρωσία θα πρέπει να βοηθήσουν για τη δημιουργία αυτών των κατάλληλων συνθήκων. οι Αμερικανοί ε, παρα, ε, διατηρεί το καθεστώς κυρώσεων. Οι κυρώσεις τώρα θα επεκταθούν και σε επιχειρηματίες και σε όσους παράγουν ε, χημικά όπλα. Οι αραβικές χώρες ανησυχούν για, την, για το ότι η, αραβική φύση του, της Συρίας ας πούμε διαβρώνεται και με μεγαλώνει η επιρροή του Ιράν, της ε, Τουρκίας και της ε, Ρωσίας. Ορισμένοι δεν θέλουν να ομαλοποιήσουν πείσουν τι ε, σχέσει του, αλλά κάποιοι όπω το Παχρέιν και τα λοιπά ε, προσπαθούν να μολυμίσουν τι σχέσει με την ε, Συρία, ανοίγουν πρεσβείε και τα λοιπά και μιλάνε για την πιθανή επιστροφή της στο στον Αραβικό Σύνδεσμο ε, όταν γίνει ας πούμε η Σύνοδος Κορυφής ε, στην Τίνιδα το Μάρτιο θα συζητηθεί το θέμα. Με βάση αυτές τις εξελίξεις εμείς ε, η θέση μας για την επιστροφή των προσφύγων, την ανοικοδόμηση και την κανονικοποίηση ε, μπορούν να έχουμε κάποιες θέσεις οι οποίες μπορούν να αμφισβητηθούν όμως. Και αυτό λοιπόν ε, σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικό να παραμείνουμε ενωμένοι και δυνατοί σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή του ψηφίσματο 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας και να μην παραδώσουμε έτσι την, ε, και εγκαταλείψουμε την επιρροή που έχουμε. Ε, εάν δεν αλλάξει η πολιτική του καθεστώτος, δεν είναι καλή τώρα φάση για την ομαλοποίηση των σχέσεων και θα είναι αναποτελεσματική κάτι τέτοιο για να αλλάξει η συμπεριφορά του καθεστώτος. Δύο λόγια για την επερχόμενη διάσκεψη για τη Συρία ε, και τι είπε ε, και τη συμμετοχή της Μογκερίνη στην σύνοδο αυτή 12 ε, με 14 ε, Μαρτίου. Θα επαναδιατρανώσουμε την ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συρία και να εξηγήσουμε γιατί δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε παραχωρήσει στο καθεστώς. Η διάσκεψη θα δείξει ότι υποστηρίζουμε τη διαδικασία του ΟΗΕ και θα χρησιμοποιήσουμε τη διάσκεψη για να εξασφαλίσουμε συνεχή ε, χρηματοδότηση για τα ανθρωπιστικά θέματα, για τους πολίτες της Συρίας και για την υποστήριξη των χωρών υποδοχής προσφύγων, σύρων προσφύγων. Θα δοθεί έμφαση στη ε, διάσκεψη για την κοινωνία των πολιτών, η οποία, όπως είπα, παίζει σημαντικό ρόλο. Ο ρόλος των γυναικών, η λογοδοσία, είναι άλλα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στη διάσκεψη. Μακρηγόρησα, θα σταματήσω εδώ. Προσβλέπω στην συζήτηση που θα ακολουθήσει και στις ερωτήσεις που θα μου υποβληθούν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φερέρ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην ε, Λίνα Κατίμπ για να μας δώσει τη δική της εκτιμήση της κατάστασης. Σας ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που με καλέσατε σήμερα το πρωί, διότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα προσπαθήσω να σας ε, δώσω μια διαφορετική εναλλακτική ε, προσέγγιση. Αποχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες και ποιος αποφελείται λοιπόν. Ακούσαμε ήδη την Έρικα ε, να αναφέρει κάποια από τα πιθανά σενάρια. Πρώτον, ISIS φυσικά είναι κάτι που ανησυχεί όλους. Ένας από τους μεγαλύτερους νικητές της αποχώρησης των Αμερικανικών δυνάμεων είναι το ISIS. Ήδη έχουν προχωρήσει από την έρημο ανάμεσα στο Ιράκ ε, και τη Συρία σε ε, Συριακό έδαφος. Οι ηγέτες λοιπόν του ISIS είναι βόρεια του Μπουκανάλ. Είναι στα βορειοανατολικά λοιπόν μια πάρα πολύ ισχυρή παρουσία του ISIS και προσπαθούν να επανενεργοποιήσουν ε, την οργάνωση. Έχουμε δει πως ε, έχουν αναλάβει μέχρι τώρα μια σειρά ε, δράσεων και δολοφονιών δημοκρατικών ε, δυνάμεων στην Συρία. Οι εντάσεις αυτές θα κλιμακωθούν περαιτέρω ε, μετά την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων, διότι δεν θα υπάρχει κανείς ε, που να μπορεί να αντισταθεί στο ISIS. Και δεν νομίζω πως ο διεθνής συνασπισμός κατά του ISIS θα μπορέσει να κάνει τίποτα χωρίς την ηγετική ικανότητα των ΗΠΑ. Υπάρχει και κάτι ε, άλλο επίσης, ε, το ποιος ε, θα επωφεληθεί. Οι αντάρτες από, από το Ιράν, ορισμένες... Ε, Ορισμένοι αντάρτε, όπω για παράδειγμα μέλη τη Χεσμολάχ, έχουν έρθει από γειτονικέ χώρε, από το Λίβανο το, και το Ιράκ. Όμω οι δυνάμει αυτές τώρα που έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι μάχες κατά του ISIS στο Ιράκ πρέπει να ε, βρουν κάτι να κάνουν. Γι' αυτό λοιπόν κοιτάζουν προς ε, τη Συρία. Εάν το ISIS επωφεληθεί τότε οι αντάρτες αυτοί θα ε, επωφεληθούν επίσης και θα βλέπουμε λοιπόν όλο ένα και περισσότερους αντάρτες που στηρίζονται από το Ιράν να πολεμούν στην ε, Συρία με το πρόσχημα της μάχης κατά του ISIS. Τώρα, τι συμβαίνει ε, στις σχέσεις μεταξύ των ανταρτών αυτών και του ISIS. Υπάρχει ε, αβεβαιότητα. Σίγουρα δεν ε, πρέπει να παραβλέπουμε την οικονομική δραστηριότητα στα σύνορα Συρίας-Ιράκ ανάμεσα σε αντάρτες που στηρίζονται από το Ιράν και το ISIS. Αυτές οι δύο οντότητες έχουν παρελθόν και τώρα που έχει νικηθεί το ISIS στο Ιράκ, έχουν πάρει αυτό που ήθελαν από τη μάχη. Έχουν πάρει εδάφη, πολιτική, πολιτικό κύρος και αυτό που μένει είναι η οικονομική διάσταση, τα οικονομικά ωφέλη. Το ISIS δεν έχει διαλυθεί. Ε, το αντίθετο έχει μετατραπεί σε μια οικονομική μαφία που δράει υπογείως και πολλοί ε, που πολέμησαν με το ISIS ως ε, μαχητές ή ως πράκτορες, τώρα είναι ε, άνθρωποι που ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ε, νόμιμες και παράνομες. Αυτό φυσικά δεν πρέπει να μας εκπλήσει, διότι τέτοια πράγματα γίνονται ε, σε εμπόλεμε ζώνες σε όλο τον κόσμο. Ε, το πότε φανταστείτε μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Πολιτειών τι θα γίνει στην περιοχή αυτή. Οι αντάρτες θα έχουν και εκείνη πρόσβαση στους ε, πόρους εκτός από το ISIS. Θα δούμε λοιπόν μία αύξηση της ε, αποσταθεροποίησης, θα δούμε περισσότερες, ε, περισσότερους ε, τέτοιους αντάρτες να εμφανίζονται και να δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Η Παραστρατιωτική λοιπόν αυτή η δραστηριότητα συνεχίζεται, αυξάνεται και πριν από μερικές μέρες έλαβε τεράστιες διαστάσεις με την δημόσια ανακοίνωση ότι στη Νότια Συρία θα γίνουν επιθέσεις κατά ε, Ιρανικών στόχων. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιρροή του Ιράν στη Συρία ολοένα και αυξάνεται. Τώρα, όπως είπε και η Έρικα, οι δυνάμει στα βορειοδυτικά όπως η HTS υποφελούνται και εκείνες από τις εξελίξεις, ε, δεδομένου ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί να ε, καταστήλει το HSDS. Ε, και μάλιστα υιοθετεί διαφορετική στάση. Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί να εξαγοράσει χρόνο έτσι ώστε να προσπαθήσει, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει, να σπρώξει το HSTS προς μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των πραγμάτων. Και για τον λόγο αυτό δεν βλέπουμε να γίνεται κάποια μάχη, να γίνονται προσπάθειες για την ε, καταπολέμηση του HSTS στην ε, Συρία. Η Τουρκία φυσικά δεν μπορεί μόνη της ε, να κάνει τίποτα, περιμένει την στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών και αυτή τη στιγμή όμως βρίσκεται η περιοχή στη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας διότι η Δύση την έχει εγκαταλείψει. Η Τουρκία λοιπόν Ελήψη στήριξη από τι Ηνωμένε Πολιτείε θα κάνει ότι μπορεί ίσα για να μπορεί να έχει ένα λόγο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να μπορεί να επηρεάσει τι εξελίξει ε, στο καθεστώ ε, τη ε, Συρία για λόγου σταθερότητα εντό Τουρκία. Φυσικά οι περιοχές στα βορειοδυτικά εξακολουθούν να είναι προβληματικές και αυτή τη στιγμή είναι το προσπάθειες για να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Αν η Τουρκία καταφέρει να σπρώξει το ε, HDS προς μια ρεαλιστική θεωρήση των ε, πραγμάτων, τότε ε, θα μπορούν να ισχυριστούν ότι έχουν ξεπεράσει την παρανομία και μπορούν να είναι υπολογίσιμοι νόμιμη πολιτική δύναμη. Οι δυνάμεις λοιπόν ε, που στηρίζονται από το Ιράν στη Συρία δεν ε, έχουν τέτοια ε, αντιμετώπιση, ακριβώς διότι υπάρχει η ρωσική στήριξη. Η συμμαχική βέβαια σχέση Ρωσίας-Συρίας είναι μία παροδική σχέση. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία προσπαθεί να βρει τόπους τρόπους αντιμετώπισης ε, του Ιράν σε Συριακό έδαφος. με στόχο να μείνουν οι δυνάμεις που στηρίζονται από το Ιράν εκτός Συρίας. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι επειδή το καθεστώς δεν μπορεί να ε, αντιμετωπίσει την ε, κατάσταση χωρίς ε, την συνδρομή της Ρωσίας. Γι' αυτό λοιπόν η Ρωσία δεν επιθυμεί το Ιράν στην περιοχή. Φυσικά Πολλέ είναι οι ενδείξεις που μας κατευθύνουν προς ε, αυτήν την ε, άποψη. Ακριβώς διότι πρώτον το Ιράν είναι μια δύναμη που ανησυχεί πάρα πολύ τις ε, Ηνωμένε Πολιτείε. Επίση, η σχέση Ρωσία και Ιράν είναι εξίσου ανησυχητική και α μην ξεχνάμε ότι οποιαδήποτε παραστρατιωτική δύναμη στηρίζεται από άλλη χώρα είναι από μόνη τη ανησυχητική είδηση. Αυτό που πρέπει να συζητηθεί είναι η παρουσία λοιπόν ε, δυνάμεων στη Συρία που στηρίζονται από το Ιράν και ε, παρά το γεγονός ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας ε, πρέπει να συνεργαστούν για το κοινό όφελος στην Συρία. Δεν υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε για ειρηνευτική διαδικασία ουσιαστικά χωρίς να υπάρξει συνεργασία. Και από ό,τι ακούω εγώ, οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εκείνες που πρέπει να κάνουν το πρώτο βήμα και να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτή τη στιγμή η Ρωσία είναι μόνη χωρίς αντίπαλο και εμεί ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαδραματίσει ένα ρόλο ε, μεσάζοντα να βοηθήσουν τις, ε, και να παροτρύνουν τις Ηνωμένε Πολιτείες ε, να κάνουν το πρώτο βήμα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πιέσουμε και να οθήσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείες προς αυτήν την κατεύθυνση προτού ε, επιδεινωθεί η κατάσταση. όσο περισσότερες περιοχές επανακαταλάβει το καθεστώς, τόσο πιο γρήγορα θα εξομαλυνθεί η κατάσταση. Χρειάζεται λοιπόν να αντιμετωπίσουμε με, με σιγουριά και αποφασιστικότητα την κατάσταση για να μην ε, εκτροχιαστεί η κατάσταση. Α στηρίξουμε την κοινωνία τη ε, συρία Είναι πάρα πολύ σημαντικό δεδομένων των περιστάσεων να μην πέσουμε στις ε, παγίδες του καθεστώτος της Συρίας προσπαθεί το καθεστώς της Συρίας να ελέγξει τα πάντα, να περνάνε όλα από εκεί έτσι ώστε να προβάλλει μια εικόνα εξομάλυνσης της ε, κατάστασης και να εκμεταλλευτεί την αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων για να ισχυριστεί πως έχει κατανικήσει το ISIS. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Ευχαριστώ ε, για αυτές τις δύο ε, παρουσιάσεις που μας έδωσαν πολλές ε, και σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα που μας απασχολεί. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να δώσω πρώτα το λόγο στην κυρία Βιλέρα. Είναι πραγματικά απογοητευτικό όλο αυτό. Όταν ε, πήγαμε στην Τουρκία, είχαμε αυτές τις συζητήσεις ε, με τις ε, ένοπλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. I, I think that when, when you talk about uh, Daesh coming back... Και ε, ακούσαμε ότι ε, οι Ιρανοί θα, θα πολεμήσουν την ε, ΝΤΑΕΣ και οι Κούρδοι θα προσπαθήσουν να προστατέψουν την περιοχή τους. Κοιτάξτε, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ αυτή η buffer zone που ευαγγελίζονται διάφοροι. Γιατί εδώ βλέπουμε ε, μάχες μεταξύ της ε, ε, Τουρκίας και των Κούρδων και αυτό βεβαίως δεν αποτελεί θετική εξέλιξη. Buffer zone έχει έννοια εάν είναι ειρηνική, αλλά εδώ δεν πρόκειται να είναι αυτή η περίπτωση. Άρα πού θα πάνε οι Κούρδοι και τι ρόλο, δηλαδή πού, θα, πού βρίσκονται οι Κούρδοι, μιλώντας για το SDF από άποψη στρατιωτική ε, τα πήγαιναν πολύ καλά στρατιωτικά απέναντι στον ISIS ε, ε, μέχρι να παρέμβει η Τουρκία και γι' αυτό ακριβώς προσπαθεί να ανασυντάξει δυνάμεις ο ISIS στην περιοχή. και φυσικά εάν το SDF δεν έχει ε, την, ε, τους, την, ε, τους να τους βοηθούν επιτόπου και αν έχουν απέναντί τους και την Τουρκία τότε πραγματικά μειώνονται οι ελπίδες των Κούρδων στην βορειοανατολική ζώνη και μπορεί να έρθει η Συρία και να πει στους Κούρδους να κάνουμε μια συμφωνία. Και αυτό δεν είναι καινούριο. Έχουμε δει περιπτώσεις όπου οι κουρδικές δυνάμεις ε, κατέλαβαν ε, θέσεις ε, από την ISIS και τις παρέδωσαν στην Συρία. Ο προβληματισμός μου είναι ότι το καθεστώς τώρα λέει δημόσια μπορείτε να πάρετε αυτονομία εάν συνεργαστείτε μαζί σας. Αλλά δεν νομίζω ότι τελικά θα επιτύχουν αυτό που θέλουν. Δηλαδή ε, χρησιμοποιούνται ως εργαλείο ε, από σχεδόν όλες τις πλευρές και δεν ξέρω αν τελικά θα κερδίσουν κάτι, αν θα τους μείνει κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κουζεκ Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Φερέρ το εξή. Ναι, βάλτε τα ακουστικά σας. Μια ερώτηση λοιπόν για την κυρία Φερέρ. Μας είπατε ότι η πολιτική θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν τροποποιήθηκε, δεν άλλαξε από το 2017 αλλά ήδη βρισκόμαστε στο 2019 και την σήμερα ημέρα ε, η Συριακή κυβέρνηση ελέγχει περίπου 90 να μην πω 95% ε, του, των εδαφών και η διπλωματική κατάσταση έχει αλλάξει ε, εξ ολοκλήρου. Θα ανοίξουν ε, και ε, πρεσβείες ενδεχομένως της Ειδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν, των Ηνωμένων Αραβικών ε, Εμμυράτων και θα ξαναγίνει δεκτή η Αραβική Δημοκρατία της ε, Συρίας ε, στην, ε, στον Αραβικό Σύνδεσμο στην επόμενη συνεδρίαση της Τινησίας. Επίσης, Ουγγαρία, Βουλγαρία, Τσεχία αναγνωρίζουν την νέα κατάσταση. Δεν νομίζετε ότι έφτασε η στιγμή να αλλάξουμε στάση και να είμαστε επιτόπου, να είμαστε παρόντες, μια και αλλάζουν οι συνθήκε και εν πάση περιπτώσει ε, σε αυτήν την ε, διαμάχη νικητής βγήκε η κυβέρνηση της ε, Συρίας. και μάλιστα μέσω και της πρέσβυρας της Τσεχίας μάθαμε ότι ε, οι κυρώσεις έχουν αρχίσει να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στον απλό λαό και εν πάση περιπτώσει μιλάμε εδώ για ε, μια πρέσβυρα και για μια πρεσβεία χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εμείς καταγγέλουμε βεβαίως παντού ε, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν συμμετέχει στην ανασυγκρότηση ε, και μας λένε ότι στηρίζουμε την πολιτική αντιπολίτευση. Και ποια είναι αυτή η πολιτική αντιπολίτευση την οποία υποστηρίζουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι στην ουσία ε, οι ομάδες που παρουσιάζονται ως ομάδες αντιπολίτευσης ε, ε, χρηματοδοτούνται από τις χώρες του κόλπου επομένως δεν είναι μια πραγματικά ανεξάρτητη αντιπολίτευση και μέχρι πότε θα, θα μείνουμε έξω από οποιαδήποτε διαδικασία ανασυγκρότησης γιατί ανασυγκρότηση οπωσδήποτε χρειάζεται στην περιοχή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομιλήτριες και ε, θα ήθελα απαντώντας σε αυτές τις ερωτήσεις να ε, κάνετε και τις καταληκτικές σας παρατηρήσεις. Ε, κυρία Φερέρ, ευχαριστούμε πολύ για τις πολύ άμεσες και ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Είπα επανειλημμένα, νομίζω, ότι δεν μπορεί κανείς να κερδίσει ειρήνη. Μπορεί να κερδίσει κανείς ένα πόλεμο, αλλά δεν μπορεί να κερδίσει την ειρήνη εάν δεν ε, ε, υπάρχει μία ε, σοβαρή, μεταβατική και απολύτως συμπεριληπτική περίοδος. Το καθεστώς οπωσδήποτε έχει μπει στην πολιτική διαδικασία και δεν βρίσκουμε κανένα λόγο να εμπλακούμε με, την, ε, το καθεστώς. Ναι, είναι γεγονός ότι κάποιες χώρες βλέπουν διαφορετικά την κατάσταση, αλλά παραμένουν ενισχύ τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ε, η ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης παραμένει. Και βεβαίως εμείς πρέπει να είμαστε ορθολογικοί, πραγματιστές, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι δυνατόν να εγκαταλείψουμε την στρατηγική μας και την συνέπεια ε, που έχουμε και την realpolitik που πρέπει να έχουμε. Αναφερθήκατε στην ε, αντιπολίτευση. Εμείς ε, μιλάμε και αναφερόμαστε στην κοινωνία των πολιτών. Έχουμε ε, την κοινωνία των πολιτών που αναπτύσσεται σε ολόκληρη την ε, Συρία και δεν ε, μιλάμε εμείς για την πολιτική αντιπολίτευση. Πρέπει να είναι σαφής ο διαχωρισμός. Δεν ξέρω εάν απάντησα στον προβληματισμό σας. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν πιστεύουμε ότι η ομαλοποίηση μπορεί να είναι κοντά σε οποιαδήποτε πολιτική διαδικασία, ενώ πολιτική διαδικασία είναι αυτή που χρειαζόμαστε εάν θέλουμε να επιτύχουμε βιώσιμη μεταβατική περίοδο στη Συρία. Thank you. I will just say... Ευχαριστώ πολύ. Το βασικό δεν είναι να φανταστούμε ότι θα πετύχουμε σταθερότητα και ασφάλεια και ειρήνη όσο ο Μπασάρα Λασάντ παραμένει στην εξουσία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη Μοσούλ για σύγκριση. Το ISIS στρατιωτικά νικήθηκε στη Μοσούλη. Αν πάτε στη Μοσούλη τώρα όμως και πήγα πέρυσι, θα δείτε ότι σε στρατόπεδα προσφύγων ε, οι γυναίκες είναι θύματα σωματεμπορίας. Ε, ως πόρνες χρησιμοποιούνται, ε, βιασμοί υπάρχουν, ο κόσμος είναι άνεργος, κάνει λαθρεμπόριο για να μπορέσει να βγάλετε προς το ΖΙΝ. Περιοχές ε, διάφορες δεν έχουν ανοικοδομηθεί. Ε, τα δυτικά είναι σε κατάσταση ερηπείων <laughs> της Μοσούλης και παρά να κυκλοφορούν γενικά στον κόσμο. Πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ταραχές είναι αποτέλεσμα κοινωνικής, οικονομικής αναταραχής και πολιτικής αναταραχής και όχι ιδεολογικής προπαγάνδας ομάδων όπως το ISIS. Με αυτό το καθεστώς του Μπασάρα Αλασάντ δεν πρόκειται να υπάρχει πραγματική και δίκαιη ανοικοδόμηση στη Συρία. Το καθεστώ θέλει να γίνει ανοικοδόμηση στι περιοχέ μόνο που υπάρχουν οι πιστοί στο καθεστώ και θέλει να τιμωρήσει όλου του υπόλοιπου. Επομένω, ο κόσμο θα παραμείνει ενδεή. Δεν θέλει οι πρόσφυγε να επιστρέψουν παρά τι δηλώσει. Το κάνει μόνο ούτω ώστε να το πιστέψουν αυτό και να πληρώσει ο κόσμο. Να πιστέψει το αφήγημα. Δεν πρόκειται να του αφήσει να έχουν αξιοπρεπή ζωή εάν σε καμία περίπτωση. Ε, επίσης θα βασίζεται σε αυτές τις πολιτοφυλακές που έχει δημιουργήσει, γιατί ο δικός του στρατός ε, δεν είναι σε καλή κατάσταση και όπως ξέρουμε και από το Ιράν και το Λίβανο, αυτή τη στιγμή έχει σε πολιτοφυλακές ε, που και δημιουργηθούν αυτές οι ελίτ, ας πούμε, σε μια οικονομία πολέμου. Είναι πολύ δύσκολο να τις ε, εξαλείψεις και η έλξη που θα ασκούν αυτές οι, πολιτι... οι πολιτοφυλακές θα είναι όλο και μεγαλύτερη γιατί έτσι θα έχεις και θα αυξηθεί ας πούμε, το κύρο σου και θα βελτιωθούν τα οικονομικά σου. Θα χρησιμοποιηθούν ε, αυτές οι... αυτά τα παράπονα του κόσμου από το ISIS ή από νέε ομάδε που θα προκύψουν. Δεν θα είναι κατά ανάγκη τζιχαντιστές και εξτρεμιστέ. Ε, μπορεί να είναι άλλοι τύποι εξτρεμιστέ, μη θρησκευόμενοι ας πούμε. Μπορεί να είναι κάτι ακόμα πιο ακραίο ας πούμε, από το ISIS που θα χρησιμοποιήσει την ε, θρησκευτική ιδεολογία επίσης. αυτά τα παράπονα οδηγούν σε αναταραχές και οι κοινωνικές και οικονομικές ε, ανισότητες ε, οδηγούν σε αναταραχές. Ε, το να αφήσουμε τους ανθρώπους φτωχούς και να μην έχουν τα προστοζήν θα οδηγήσει και αυτό σε αναταραχές. Επίσης, δεν μιλάμε στην πραγματικότητα για ένα κυρίαρχο στρατιωτικό κράτος υπό τον Μπασάρα, Λασάντα. Στηρίζεται από τη Ρωσία. Ε, είναι για ένα συναλλακτικό κράτος. Ε, το ε, υπάρχει ένα σχετικό έγγραφο που έχουμε δημοσιεύσει από το Chatham House και μπορείτε να δείτε τι πιστεύουμε σε αυτό το έγγραφο. το να πιστεύουμε ότι κέρδισε το καθεστώς είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί έχουμε όλε αυτέ τι πολιτοφυλακέ που ανακύπτουν, α πούμε, που είναι Σουνίτε ή και άλλες πέρα από το ISIS. Ε, και εμεί μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη είμαστε οι πιο κοντινοί δυτικοί γείτονε τη Συρία και θα επηρεαστούμε είτε μα αρέσει είτε όχι. Προσεκτικά λοιπόν πρέπει να προχωρήσουμε ε, και για να δούμε ας πούμε τι θα επενδύσουμε. Ό,τι επενδύσουμε με μεγάλη προσοχή να το επενδύσουμε στη Συρία. Ναι, δεν απάντησα την ερώτηση που αφορούσε τις κυρώσεις και για να απαντήσω φυσικά και μας ανησυχεί πάρα πολύ το ότι οι κυρώσεις δεν θα έχουν επιπτώσει σε εκείνους ε, ε, που ε, έχουν ως στόχο πολίτες απλούς, άμαχο πληθυσμό. Φυσικά και υπάρχουν εξαιρέσεις για ιατρικές προμήθειες, φάρμακα κτλ. Αλλά είναι όντως κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους ε, προσκεκλημένους μας για τις πολύ σημαντικές ε, λεπτομερείς συνεισφορές σας σήμερα. Πράγματι, το έγγραφο στο οποίο αναφέρεστε από το Chatham House είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω πως οφείλουμε όλοι να το διαβάσουμε. Ε, φυσικά και είναι λοιπόν πολύ σημαντικά τα στοιχεία που περιέχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα παρακολουθούμε λοιπόν τις ε, εξελίξεις στην περιοχή με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. So, thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την ε, κυρία Μούντι που μου έδωσε την ε, Προεδρία. Να σας καλωσορίσω όλους στην Συζήτηση για το σημείο 7 από κοινού με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων πρόκειται για τα αλλαγή απόψεων σχετικά με την κατάσταση της ασφάλειας στο Κωσυφοπαίδιο. Νομίζω πως είναι πολύ επίκαιρη η συζήτηση αυτή, διότι δύο μήνες ε, πριν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με την ανακοίνωση τη Κομισιόν, ε, σύμφωνα με την οποία χρειάζεται περισσότερη πρόοδο στο κοσυφοπαίδιο αναφορικά με την δικαστική και πολιτική συνεργασία. Από τότε έχουμε παρατηρήσει αυξημένε εντάσει στην περιοχή. Το κοσυφοπαίδιο προσπαθεί να δημιουργήσει είναι φυσικές εξελίξεις αυτές όταν προσπαθεί ε, να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτο. όμως υπάρχουν παραβιάσεις διεθνών συμβάσεων. Γι' αυτό λοιπόν ε, με χαρά μας καλωσορίζουμε σήμερα διακεκριμένους προσκεκλημένους ψηλόβαθμου ε, αξιωματούχους για να μας ενημερώσουν. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω τους εμπειρογνώμονές μας, οι οποίοι φτάνουν. Έχω Ήδη δει κάποιους ένστολους να έρχονται. Α, εδώ. Thank you So Έφτασαν λοιπόν όλοι οι προσκεκλημένοι μας, όπως βλέπετε, και θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω και να παρουσιάσω τους ε, προσκεκλημένους. Ε, πρώτα η κυρία Αννα Μαρία Μπούρα, πρόεδρος ε, της Ομάδας Εργασίας του Συμβουλίου για την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και σύμβουλος για το ε, με αυτό. Καλώς ορίσατε. Μετά ο David Κάλεν, προϊστάμενος τμήματο ε, για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονία και το Κωσυφοπέδιο από την Γενική Διεύθυνση ΝΙΑΡ της ε, Κομισιόν. Ήσασταν εδώ και την Δευτέρα το απόγευμα, οπότε σας έχουμε συχνά εδώ. Καλώς ήρθατε και τον υποστράτηγο Λορέντζο Νταντάριο, διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων στο Κωσυφοπέδιο. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Χωρίς καθυστέρηση λοιπόν, θα δώσω το λόγο πάλι στην Claire Moody. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ πολύ σύντομα θα κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια. Και φυσικά θα αρχίσω λέγοντας ότι όταν συζητάμε την κατάσταση ασφάλεια στο Κωσυφοπαίδιο πρέπει να τονίσουμε ότι η διατήρηση της ειρήνη είναι πάρα πολύ σημαντική προϋπόθεση για τις ε, σχέσεις σερβία και Κωσυφοπαιδίου και για την ε, προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσθέσω επίσης κάποια ε, σχόλια τα οποία ίσως πυροδοτήσουν τη συζήτηση. Υπάρχουν πολλαπλοί παράγοντες που ε, μας οδηγούν σε ανησυχία για κλιμάκωση της κατάστασης. Πέρυσι παρατηρήθηκε μία με μεταλλαγή ε, της ε, στρατιωτικής δύναμης του Κωσυφοπεδίου σε επαγγελματικό στρατό και αυτό έχει δημιουργήσει εντάσεις ανάμεσα στη Σερβία και το Κωσυφοπέδιο. Η K4 λοιπόν πώς εκτιμά τον ε, κίνδυνο που ενδεχομένω δημιουργείται από αυτήν την αλλαγή. Επίσης η εντολή του στρατού του Κωσοφοπεδίου θα πρέπει να αλλάξει μόνο σταδιακά μέσω μιας ομαλής διαδικασίας και κατόπιν δημιουργίας συντάγματος του Κωσοφοπεδίου το κοσυφοπαίδιο πρέπει να συνεχίσει να τηρεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις σχετικά με, τις, με τους διακανονισμούς για την ασφάλεια στην περιοχή. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα την άποψη των ε, συναδέλφων καθώς και τις εκτιμήσεις σας ε, για το αν αυτό ε, πραγματοποιείται. Επίσης, η εντολή της ΚΕΙΦΟΡ στο Κωσυφοπέδιο που οφείλει να διασφαλίσει ασφάλεια και ειρήνη στην περιοχή έτσι ώστε να εξελιχθούν οι συζητήσεις στο Φελιγράδι. Θα πρέπει λοιπόν να συνεισφέρουμε στην αποτροπή της εμφάνισης νέων απειλών. Κατόπιν ε, αυτών των σχολείων λοιπόν θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στην κυρία Μπούρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με μια σύντομη εισαγωγή σχετικά με το ε, υπόβαθρο της ε, κατάστασης. Και ο συναδελφός μου, Ντέιβιντ, είμαι σίγουρος, σίγουρη πώς θα συμπληρώσει αυτά που θα σας πω. Ε, αν με ρωτούσατε λοιπόν πώς ε, είναι η κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο θα την χαρακτήριζα ήρεμη αλλά εύθραυστη. Υπάρχει μια πολιτική πόλωση εντονότατη, υπάρχει ένας κυβερνητικός συνασπισμός ο οποίος είναι διχασμένος στο εσωτερικό του και οι, οι λόγοι του διχασμού είναι πρώτον η έλλειψη πολιτικού διαλόγου. Έπειτα υπάρχει ένας κατακαιρματισμός της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε υψηλές εντάσεις στη δημοκρατική διαδικασία και εμείς όμως προσπαθούμε μέσω, στη μέση όλης αυτής της κατάστασης να συνεχίσουμε το έργο μας. Τώρα, πώς εκτιμούμε εμείς τον κίνδυνο κλιμάκωσης και την τήρηση των δεσμεύσεων από το κοσυφοπαίδιο. Εμείς καταρχάς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να παραμείνει ε, ειρήνη στην ε, περιοχή. Προσπαθούμε καταρχά να συνεργαστούμε μαζί του για την εξομάλυνση των σχέσεων Κοσμοπεδίου Σερβία. Προσπαθούμε να ε, συνομιλούμε και με την κυβέρνηση του Κοσμοπεδίου αλλά και με δυνάμει αντιπολίτευση και έπειτα προσπαθούμε να του βοηθήσουμε έτσι ώστε να εισέλθουν σε ε, τροχιά ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια πραγματικά δημοκρατική ευρωπαϊκή τροχιά. Η διαδικασία βέβαια ε, προσχώρηση ε, είναι αρκετά απογοητευτική για το κοσυφοπαίδιο. Είχαν προσδοκίες οι οποίε παρέμειναν ανεκπλήρωτες και αυτό έχει πλήξει την αξιοπιστία μας. Αυτό που προσπαθούμε δηλαδή να επιτύχουμε στο, στη χώρα. Πέρα από τις πολιτικές όμως προκλήσεις υπάρχουν και νέα προβλήματα. Ίσως έχετε ακούσει για τους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου που ξεκίνησαν τον Νοέμβριο, άρχισαν με 15% και προχώρησαν στο 100% και αυτό έχει οδηγήσει στην αύξηση των εντάσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες αλλά και ε, εντός κοινοβουλίου ε, του Κωσυφοπεδίου έχουν λοιπόν αυξηθεί εντάσεις και με τους διεθνείς εταίρους πέραν ε, των εσωτερικών εντάσεων και η αντιπολίτευση ήταν σαφέστατη, αναμένει από την κυβέρνηση να ανακαλέσει το μέτρο αυτό διότι παραβιάζει και την ε, ε, ΕΖΕΣ και άλλες διεθνείς συνθήκες και δυσχεραίνει τις την εξομάλυνση των, ε, σχέσεων, των διεθνών σχέσεων. Αυτό έχει προκαλέσει επίσης διάφορες διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις στα βόρεια του Κωσυφοπεδίου, όμως μέχρι τώρα δεν έχουμε οδηγηθεί σε ε, κλιμάκωση της ε, βίας. Όμως ε, υπάρχουν καθημερινές διαδηλώσεις στο βόρειο Κωσυφοπέδιο από, όλες, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος λοιπόν να εκτροχιαστεί η κατάσταση στη βία. Επίσης, η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα επιβολής αντισταθμιστικών ε, μέτρων για την μετάβαση προς μια βελτιωμένη επικοινωνία μεταξύ των ε, δύο κοινοτήτων. Ε, η εκτίμησή μας είναι ότι αυτή η μετάφαση θα πρέπει να γίνει με τρόπο σταδιακό και χωρίς ε, αποκλισμούς Και Θεωρούμε πως η εφαρμογή των μέτρων αυτών θα πρέπει να γίνει με εξίσου ομαλό τρόπο. Είμαστε απόλυτα εναρμονισμένοι με τον ΝΑΤΟ σε αυτό το θέμα. Βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή και συνεργαζόμαστε στενά. Η παρουσία μας είναι έντονα ορατή στην περιοχή και θα συνεχίσουμε και με το διάλογο και με την προσπάθειά μας να επικοινωνήσουμε και να είμαστε συνεχοχοί επαφή με τις αρχές στην Πρίστινα, να γίνονται έλεγχοι για την ε, τήρηση του κράτους ε, δικαίου. Η EULEX βρίσκεται επί τόπου. Υπάρχει νέα εντολή για την ε, ομάδα αυτή, η οποία θα συνεχίσει μέχρι το 2020 αποτελείται από 500 περίπου άτομα και ε, πολίτες του Κωσίφοπεδίου αλλά και ε, διεθνείς ε, δυνάμεις. Το ΝΑΤΟ επίσης είναι ο τρίτος εγγυητής ασφάλειας στην περιοχή και στο πλαίσιο αυτό εμείς συνεχίζουμε να ε, κάνουμε προσπάθειες προς ε, την βελτίωση της ε, ασφάλειας. Όμως, για να εξασφαλιστεί ουσιαστική πρόοδος ε, και ειρήνη στο κοσυφοπαίδιο, πρέπει πρώτον να εξομαλυνθούν οι σχέσεις, δεύτερον να βελτιωθεί ο διάλογος και τρίτον να τεθούν κάποια θέματα στην ημερήσια διάταξη. Θα σταματήσω εδώ και θα σας δώσω το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τον κύριο Κάλαν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπε μόλις η κυρία Μπούρα, πάντως συμφωνώ με την αξιολόγηση που έχει κάνει. Η κατάσταση είναι ήρεμη, αλλά ε, ιδιαίτερα εύθραυστη. Βλέπουμε επίσης ε, και στον Βορρά να είναι ιδιαίτερα δύσκολη η κατάσταση. Τις ε, τελευταίες εβδομάδες είχαμε αρκετά προκλητικά ζητήματα και δύσκολα, όπως ας πούμε το θέμα και των δασμών. Αλλά πρέπει να πούμε ότι το θέμα των δασμών κατά την άποψή μας είναι ε, ε, μέτρο ε, που βεβαίως αντιτίθεται και στο πνεύμα του DSAA και της ΣΕΦΤΑ είναι κάτι το οποίο ε, μελετά πολύ προσεκτικά ο Επίτροπος ε, Χάν. Ε, δύο φορές πήγε στην Πρίστινα και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν εκεί και παρακολουθεί στενά το θέμα. Αλλά ας δούμε το ευρύτερο, την ευρύτερη εικόνα. Τα βασικά νομικά έγγραφα τα οποία μας οδηγούν είναι τα κείμενα του SAA. Αυτά μας καθοδηγούν, καθώς επίσης και η στρατηγική της Κομισιόν για τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, πρώτα απ' όλα εμείς ε, ε, προσπαθούμε να πούμε στις αρχές ότι θα πρέπει να ενστερνιστούν κάποιες από τις βασικές αρχές και βάσει και της ULEX που είναι εκεί καθώς επίσης και βάσει της αναθεωρημένης εντολής της ULEX βεβαίως μας ενδιαφέρει η εφαρμογή των στοιχείων να γίνεται με ομαλό τρόπο έτσι ώστε να γίνει σωστά επίσης υποστηρίζουμε τον διάλογο ε, μέσω ε, προηγουμένων ε, συμφωνιών και στοιχείων που έχουν ήδη συμφωνηθεί ε, και βεβαίως μας ενδιαφέρει πάρα πολύ η ασφάλεια σε όλα τα Δυτικά Βαλκάνια. Ε, η ασφάλεια των συνόρων συνεπάγεται, ε, διορθώνω, η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέει και από την ασφάλεια των συνόρων. Και βεβαίως αυτό σημαίνει ότι βάσει των αξιών μας και των κεκτημένων μας θα πρέπει να ακολουθηθούν ε, κάποιες ε, οδοί από την ε, χώρα. Το κράτος δικαίου συμπεριλαμβάνει και την ασφάλεια και εμείς είμαστε απόλυτα συνδεδεμένοι και προσιλωμένοι μάλλον στο κράτος δικαίου. Εάν δει κανείς τα στοιχεία όσον αφορά τα στοιχεία 54,6 εκατομμύρια από το 14 ε, μέχρι το 18 και άλλα 35 για την επόμενη περίοδο 18 18 με 20. Ε, και επομένως αυτό δείχνει και το ενδιαφέρον το οποίο δίνουμε, αποδίδουμε σε αυτήν την κατάσταση. Θέλουμε ε, να βοηθήσουμε το κοσυφοπέδιο να ενδυναμώσει τις ε, αρχές δικαίου και το, το σύνταγμά του και να παρέμβουμε οπουδήποτε χρειάζεται. Συνεργαζόμαστε στενά με όλους τους εταίρους εθνικούς και διεθνικούς. Υπάρχουν και κάποια προβλήματα όμως τα οποία σχετίζονται με την αστάθεια και την ασφάλεια. Πρώτα απ' όλα ε, η αστυνομία του Κωσυφοπεδίου ε, έχουν ε, κάποιες δυνάμεις με σωστή εντολή, με καλή προετοιμασία και κατάρτιση. Εμείς τους βοηθούμε με συγκεκριμένη χρηματοδότηση έτσι ώστε να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή αστυνομία. Επίσης, η τα τελωνία κάνουν καλή δουλειά όσον αφορά τον εντοπισμό μικρών όπλων. Δουλεύουν επίσης και βάση της μεθοδολογίας, της πιο τελευταίας μεθοδολογίας ε, αξιολόγησης ε, απειλής. Ε, και βεβαίως το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό, κυρίως όσον αφορά οργανωμένο έγκλημα και διαφθορά. Second area I want... Ε, υπάρχουν και άλλα στοιχεία όπως είναι ας πούμε η, ε, ε, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και η αποτροπή βιαίων εξερμιστικών πράξεων. Εμείς βεβαίως θέλουμε να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον κίνδυνο ενδεχόμενης τρομοκρατικής επεν επέμβασης. Ε, από το 2014 είχαμε πληροφορίες και για ε, περάσματα συνόρων από ύποπτα ε, άτομα, αλλά πάντως από το 2014 και μετά δεν υπάρχει ανοιχνεύση τέτοιων μαχητών. Ε, η ασφάλεια ε, και το δικαστικό ε, τμήμα στο Κωσυφοπαίδιο. Εκεί καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες έτσι ώστε οι επαναπατρισμένοι μαχητές να μην αποτελέσουν κίνδυνο για την κοινωνία. Οι προσπάθειες συνεχίζουν και μάλιστα προοδεύουν. Τέλος, όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα και καταπολέμηση αυτού, εδώ έχουμε σημαντικά προβλήματα στο κοσυφοπαίδιο και πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν επιπλέον μέτρα έτσι ώστε να μην να διασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική ανάμειξη ε, στις ε, ε, προσπάθειες της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Πέρασε στην Ολομέλεια πρόσφατα η αλλαγή του ποινικού κώδικα καθώς επίσης και στοιχεία όπως ας πούμε το πάγωμα και η κατάσχεση περιουσιών ε, οι διαδικασίες ε, ποθενέσχες, δήλωση εισοδημάτων κλπ. Όλα αυτά είναι θετικά. Συχνά η κατάσταση όμως ε, στο κοσυφοπέδιο επισκιάζεται από ένα-δύο μεμονωμένα περιστατικά, ενώ γίνεται δουλειά σε γενικές γραμμές. Θα πρέπει οπωσδήποτε όμως να διασφαλίσουμε ότι αυτή η καλή νομοθεσία θα ακολουθηθεί από σωστή εφαρμογή ε, το θέμα της ε, κατάσχεσης ε, των περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται πάντοτε και χωρίς καμία εξαίρεση. Ολοκληρώνοντας να πω κυρία Πρόεδρε και κύριε Πρόεδρε ότι θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ε, το κοσυφοπαίδιο σε όλους τους τομείς ε, της ασφάλειας, της σταθερότητας και της εφαρμογής του κράτους δικαίου. Ωστόσο θα πρέπει να έχουμε ε, και εστιασμένη δέσμευση από πλευρά των αρχών του κοσυφοπεδίου έτσι ώστε και το Κωσυφοπαίδιο να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη και να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις που έχει ήδη αναλάβει και τις υποχρεώσεις που έχει ήδη υπογράψει. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν εμείς θα θέλαμε άρση ε, των εμπορικών μέτρων, επιβολής δασμών κλπ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Τελευταίες παρατηρήσεις. Ο υποστράτηγος ε, ε, Λορέντζο Νταντάριο. Μακάρι να σας είχα ακούσει καλύτερα. Κάντε λάθος τον τίτλο μου, δεν πειράζει. Με είπατε αντιστράτηγο, είμαι υποστράτηγος. Ε, είμαι ο διοικητής των δυνάμεων ε, εδώ και λίγους μήνες, ανέλαβα τέλη Νοεμβρίου. Όπως ξέρετε το ψήφισμα 1244 του 1999 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ε, θεωρεί ότι η δύναμη K4 είναι υπεύθυνη δύναμη για την ασφάλεια α, του Κόσοβο. Ως διοικητής του Κοσφοπεδίου έχω στρατιωτική ιδιότητα, δεν ασχολούμαι πολιτική, αλλά ε, βλέπω τις συνέπειες της πολιτικής ε, στο Κοσφοπέδιο. Το πιο σημαντικό ε, αυτό που διαμορφώνει το, δικό μου πεδίο αρμοδιοτήτων είναι ότι ένα επιθετικό ε, πολιτικό περιβάλλον ε, μας επηρεάζει. Δεν είναι η πρώτη μου αποστολή στο Κοσφοπέδιο. Έχω, ήμουν στην αρχική αποστολή. Ε, ήδη ε, 28 κράτη συνεισφέρουν και περίπου 3.600 στρατιώτες και ε, μη στρατιώτες. Ε, δουλεύουμε πολύ, πολύ με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την τον εκπρόσωπό σας. Ε, βλεπόμαστε μία φορά τη βδομάδα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας για να συντονιστούμε και νομίζω ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να δούμε τι θα, πώς θα τελεσφορήσει η αποστολή μας. Ε, συμφωνώ απόλυτα με τις αξιολογίες σας για τα διάφορα στοιχεία. Το μόνο που θέλω να σας πω είναι ότι ε, η Ειδική Συνόδος άρχισε την, να κάνει συνεντεύξεις με κόσμο. Το ειδικό δικαστήριο μάλλον. Και θέλω να σας πω ότι ο πληθυσμός είναι πολύ ανήσυχος, ειδικά οι νέοι ε, είναι πολύ απογοητευμένοι. Ε, ειδικά για το θέμα της απελευθέρωσης από την υποχρέωση θεωρήσεων για την ε, επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προκλητικές ε, δηλώσεις και οι ρητορίες ε, χρησιμοποιούνται για εσωτερική κατανάλωση, για συγκεκριμένους ε, ψηφοφόρους και προκαλούν αυτή την τον πολιτικό κατακαιρματισμό για τον οποίο μιλήσατε. Κανένας δεν θέλει να προκαλέσει εκ ε, την επιστροφή στο κλίμα του 2004 με βίες ανταλλαγές ας πούμε. Αυτό που με ανησυχεί είναι αυτή η έφλεκτη ατμόσφαιρα μπορεί να δημιουργήσει το κατάλληλο περιβάλλον για μεμονωμένα περιστατικά που έχουμε σήμερα, τα οποία αύριο μεθαύριο θα οδηγήσουν σε αλυσιδωτές αντιδράσεις. Αυτό δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Ορισμένα ΜΜΕ ε, δημιουργούν, μιλάνε για, με έναν τρόπο για τις ειδήσει. Ε, και δημιουργούν ένα τέτοιο κλίμα, ας πούμε, που συνεισφέρει σε αυτήν την κατάσταση. Φυσικά υπάρχουν πολλά παράπονα, ε, δυσφορία σε συνδυασμό με την ε, απογοητεύση των νέων, την οικονομική κατάσταση του κόσμου κτλ. Ε, μπορεί να οδηγήσουν σε κάποια έτσι, επεισόδια. μαζί με τις άλλες ε, διεθνείς οργανώσεις, ειδικά την Ευρωπαϊκή Ένωση, διερωτόμαστε πού μπορεί να οδηγήσουν αυτές οι δηλώσεις, αυτές οι ρητορίες και ξέρουμε ότι δεν βοηθούν. Η K4 παίζει σημαντικό ρόλο για την ασφάλεια και πιστεύουμε ότι η ασφάλεια είναι μια προϋπόθεση εκ των όνου αν και όχι ικανή για να οδηγήσει σε διάλογο. Τους προηγούμενους μήνες ο προκάτοχός μου και εγώ σε συμφωνία με τους ανωτέρους μας υιοθετήσαμε μια δραστήρια στάση για να εξασφαλίσουμε ότι όταν προβλέπουμε εντάσεις μετά την ίσπραξη των φόρων, ας πούμε, Φερρυπίνη, στα βόρεια του Κοσφοπεδίου, υπήρχαν ειρηνικέ διαπραγματεύσει από διάφορε κατηγορίε ε, πολιτών και εμεί παρακολουθούσαμε εκ του σύνεγγυ. Ε, είχαμε ε, ομάδε αναγνώριση, ε, τι οποίε είχαμε αναπτύξει πριν από την ε, ε, πορεία, ας πούμε, και διαδήλωση, ούτως ώστε να προλάβουμε τις εκτροπές το κάναμε αυτό, ούτως ώστε να είμαστε επιτόπου, να μπορούμε να παρέμβουμε, αν χρειαστεί, ε, άμεσα. Και η Γιούλεξ σε μια δεύτερη φάση, σε δεύτερο χρόνο. Κυρίω όμως, να δώσουμε και μια άνεση, μια βεβαιότητα στην αστυνομία. αστυνομία. Φανταστείτε ένα νέο ε, αστυνομικό λοχείο, ας πούμε, ε, στα βόρεια της Μητρόβιτσα, ας πούμε. που έχει, ας πούμε, εντάξει, έρχεται σε σε επαφή ας πούμε με άλλους ε, ας πούμε ε, καταλαβαίνετε ότι αισθάνεται το βάρος και της ευθύνης και την πίεση. Προσπαθούμε να αποτρέψουμε το να ξεσπάσουν επεισόδια και να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει καμία πρόθεση για δημιουργία βίας. Αλλά επειδή υπήρχε αυτό το κλίμα, ας πούμε, το οποίο ήταν κατάλληλο ε, και θα μπορούσε να υποθάλψει τέτοιες, τέτοια βία περιστατικά, ε, τέτοια βία επεισόδια. Από το Δεκέμβριο μέχρι σήμερα, ε, σε ό,τι αφορά το δυναμικό της και η δεν έχει αλλάξει τίποτα. Πρόκειται για ένα δεκαετές σχέδιο ε, το δυναμικό μας θα αυξηθεί βαθμιαία μέσω ενός σχεδίου που έχουμε ετοιμάσει. Και το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πει ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο που δημιουργήθηκε αυτό το σχέδιο, με το πώς πέρασαν ε, διάφοροι νόμοι χωρίς διαβούλευση. Ε, δεν, δεν μας άρεσε και ο χρονισμός, αλλά αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Και Όλα αυτά συμβαίνουν με ένα ε, συγκεκριμένο βήμα ε, μέσα σε πλαίσιο ειρήνης. Αλλά παρόλα αυτά και στη Σερβία και στο Κοσμοπέδιο υπάρχει ένα στρατός που υποτίθεται είναι το εργαλείο για να στηρίξει την κυριαρχία και αυτό μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Ε, αν το KSF στο βορρά θεωρηθεί ότι είναι επικίνδυνο, ε, μπορεί να προκαλέσει εντάσεις κτλ. Εμείς επαγρυπνούμε γιατί Καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα κλίμα το οποίο δημιουργεί ο στρατός, ένα κλίμα το οποίο δεν υπήρχε πριν. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα αποφασίσει αυτή τη βδομάδα τη θέση του για το KSF. Επιθυμούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να έχουν ενιαίο μέτωπο απέναντι στο KSF και γενικά για αυτό το θέμα. Ε, δεν προβλέπεται να υπάρξει ρήγμα. Πρέπει να στείλουμε ένα ενιαίο μήνυμα, αλληλεγγύη, αλληλέγγυο μήνυμα Κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολούμαι με το κοσμοπέδιο. Ε, από τη στιγμή που έφτασα, αισθάνομαι ότι το K4 ε, είναι έτοιμο πόλεμο, μπορεί να παρέμβει ε, και οι δύο πλευρές το θεωρούν χρήσιμο, χρήσιμη δύναμη. Είναι μια στρατιωτική παρουσία ε, με σαφέ σχέδιο, με σαφή ιεραρχία. και πολυεθνικό χαρακτήρα, άρα ευελιξία τη δυνατότητα ανταπόκρισης, απόκρισης μάλλον, ε, για οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε περιοχή. Συνεργαζόμαστε με πολλούς φορείς και θεσμούς του κοσφοπεδίου, με τις άλλες διεθνείς οργανώσεις και προφανώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε συνομιλίες με τον Σερβικό στρατό και αυτό είναι πολύ σημαντικό Έχουμε ανταλλαγές απόψεων με το Σερβικό Υπουργείο Άμυνας και το γεγονός αυτό ε, βοηθάει τους Κωσοβάρους να μην δημιουργούν λάθος αντιλήψεις μέσω ας πούμε της δικής μας διαμεσολάβησης. Ε, φέτος θα γιορταστεί η 20η επέτειος από την έναρξη της αποστολής του K4 στο Κωσφοπέδιο και πιστεύουμε ότι θα είναι κατάλληλη στιγμή για να δούμε τι πρόσφεραν αυτά τα 28 κράτη σήμερα, ε, γιατί υπήρχαν πολύ περισσότερα και άλλα έθνη που συμμετείχαν, στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους. Υπάρχουν ε, κάποιοι οι οποίοι έχουν το βλέμμα στραμμένο στο παρελθόν. Το θέμα είναι να στρεφόμαστε προς το μέλλον τις αλλαγές που θα γίνουν κτλ. Φτάνουν αυτά. Μπορώ να σας απαντήσω σε ερωτήσεις και σε ευχαριστώ που μας προσκαλέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Έχουν ήδη ζητήσει κάποιοι συνάδελφοι το λόγο, αλλά πρώτος θα ξεκινήσει ο κύριος Μακάλιστερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μούντι. Έχω δύο ερωτήσεις. Μία προς τους εκπροσώπους της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλη μία ε, προς τον ε, Ιταλό υποστράτηγο. Πρώτη ερώτηση. Νομίζω πως συμφωνούμε όλοι ότι οι δασμοί που έχουν απευληθεί από τους Κωσοβάρους είναι απαράδεκτοι. Είναι ξεκάθαρη παραβίαση της συμφωνίας ΣΕΦΤΑ. Αλλά με όποιον συνομιλώ υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση. Είναι πράγματι απαράδεκτη κατάσταση, όμως οι δασμοί υπάρχουν. Τι μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να πείσουμε το κοσυφοπέδιο ότι αυτή είναι λάθος κίνηση και τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να αυξήσουμε την πίεση προς το κοσυφοπέδιο. Είναι κάπως προκλητική η ερώτησή μου. Ε, αυτό διότι κάνουμε τόσο πολλά για εκείνους ε, και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε και κάτι σε ανταπόδοση. Ή μήπως ζητάμε πάρα πολλά. Προσπαθώ λοιπόν να καταλάβω τι έχουμε κάνει και τι πρέπει να κάνουμε, τι πρόκειται να κάνουμε, διότι η κατάσταση ιδιαίτερα ανάμεσα στους ε, Σέρβους στο Βόρειο Κωσυφοπαίδιο είναι αρκετά άσχημη. Υπάρχει μεγάλος ε, εκνευρισμός. Ήμουν εκεί πέρυσι το Νοέμβριο, πήγαμε και στο Βελιγράδι και στην Πρίστινα και σταματήσαμε στη Μητροβίτσα. Έτσι κάναμε έναν ωραίο περίπατο στην πόλη και στις διόχθες του ποταμού. Είχα αρκετέ ε, πολύ φιλικέ συζητήσει πάνω στη γέφυρα με Ιταλού καραμπινιέρου και με πολίτε ε, και μάλιστα παρατήρησα ότι χάρηκαν πάρα πολύ που συνάντησαν ε, αξιωματούχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να ρωτήσω τον υποστράτηγο Νταντάριο εάν θεωρεί ότι Ιδιαίτερα για τη σερβική μειονότητα στο Κωσυφοπαίδιο, πως υπάρχει κάποια βελτίωση στην κατάσταση ασφαλείας στο βόρειο Κωσυφοπαίδιο και τι γίνεται με τον ε, σερβικό θύλακα στο νότιο Κωσυφοπαίδιο. Είχα συνομιλίες με εκπροσώπους της σερβικής κοινότητας και ε, στις δύο πλευρές. Και επίσης θα σταλεί και μία αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων από τις 27 Φεβρουαρίου μέχρι τις 2 Μαρτίου στην ε, Πρίστινα και σκοπεύουμε να περάσουμε μισή μέρα στη Μητροβίτσα για να συναντήσουμε εκπροσώπους της αλβανικής και της σερβικής κοινότητας του Κοσφοπεδίου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πίτσουλα, θα θέλατε κι εσείς να κάνετε κάποια ερώτηση. Παρακαλώ, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας και για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες που μας δώσατε. Πράγματι είναι πολύ δύσκολο να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι πολίτες του Κωσυφοπεδίου χρειάζονται θεωρήσεις για να μπορούν να ταξιδέψουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι το κοσυφοπαίδιο έχει ε, ότι το κοσυφοπαίδιο πληρεί σχεδόν όλες τις προϋποθέσεις ε, για να ταξιδεύει κανείς από εκεί χωρίς θεώρηση. Οι πολίτες πρέπει λοιπόν ε, να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα και αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, όχι μόνο εμείς αλλά και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Επίσης να αναφέρω ε, πως ε, έχουμε χάσει αρκετές ευκαιρίες. Δηλαδή, τι εννοώ, η περσινή χρονιά ξεκίνησε πάρα πολύ καλά. Είχαν γίνει πολλές θετικές ενέργειες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για παράδειγμα η αξιόπιστη στρατηγική διεύρυνση, η οποία πήγε μπροστά όλη την ε, περιοχή των δυτικών αυτών Βαλκανίων, όμως μετά την σύνοδο στην ε, Σόφια τον Ιούνιο ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων ε, υπήρξαν πολλοί δισταγμοί και μείναμε πολύ πίσω ως προς την πρόοδο. Αυτό οδήγησε στην αύξηση των εντάσεων, όπως είπατε και εσείς, στην περιοχή αυτή και είχαμε ως αποτέλεσμα εισαγωγή δασμών στη Σερβία και τη Βοσνία Ριζεγοβίνη αυτή η αγανάκτηση δεν είναι αισθητή μόνο στο Κωσυφοπαίδιο αλλά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να σας πω. Πολλοί συνάδελφοί μου, ευρωβουλευτές, επένδυσαν, προσπάθησαν να βοηθήσουν το Κωσυφοπαίδιο να ε, καταφέρει να φτάσει μέχρι εδώ, όμως το μέλλον δεν είναι τόσο λαμπρό. Είμαστε δύο μήνες περίπου πριν τις ευρωεκλογές και Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, δεν βλέπω περιθώρια βελτίωσης ή ε, ουσιαστικής ή μικρής έστω. Δεν βλέπω κάποια ευρωπαϊκή προοπτική ικανή να μειώσει τις ε, εντάσεις. Αλλά αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι ότι δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα μείωση ε, της ένταση εντό κοσμοπεδίου. Η εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να παραμένει μεγάλη, όμως ε, αυτό αλλάζει, ξέρετε, πολύ γρήγορα. Ερώτηση λοιπόν. Δεν άκουσα μέχρι τώρα από εσάς κάποια άποψη για το τι γίνεται με την επιρροή ξένων φορέων και ε, αναφέρομαι σε ορισμένες περιπτώσεις ε, από ε, απαγωγών Τούρκων ε, πολιτών που έγιναν με τη βοήθεια της αστυνομίας ή των ε, υπηρεσιών πληροφοριών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει μία έντονη παρουσία, διότι διαφορετικά αυτά τα φαινόμενα θα ε, παρατηρούνται όλο και συχνότερα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κούκαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες που μας δώσετε. Νομίζω ότι χρησιμοποιούμε υπερβολικά διπλωματική γλώσσα. Η ερώτησή σας είναι πολύ σωστή. Είπατε και οι δύο ότι η κατάσταση στο κοσυφοπαίδιο είναι ήρεμη αλλά ε, εύθραυστη. Εγώ τη βλέπω εντονή και εν δυνάμει εκρηκτική. Μακάρι να είσαστε εσείς ε, σωστοί και εγώ λάθος, αλλά μέχρι τώρα δεν μας έχετε πείσει. Μιλάτε για βασικά θέματα, την αύξηση κατά 100% των δασμών. Ο Τονίν έχει δίκιο. Όλοι τους το λένε. Και αυτοί λένε ναι σας ακούμε, σας ακούμε, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κατάσταση. Όσον αφορά το, τον στρατό. Όλοι τους το είπανε, με πρώτον το Στόλτεμπρεκ να μην το κάνουνε, αλλά προχωράνε. Πέρασε και ο νόμος από το Κοινοβούλιο, ε, ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός θα έχουν υπογράψει όλα, επομένως τι θα γίνει μετά. Ακόμα ελπίζουμε ότι θα κάνουν κάτι άλλο. Έχουμε επιχειρήματα ή μονάχα την ελπίδα έχουμε σαν κύριο επιχείρημα ότι θα ελπίσουμε δεν θα το κάνουνε. Μακάρι να είχα λάθος, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει πολύ σοβαρά να λάβουμε υπόψη όλα τα θέματα αυτά. Δεν θέλω να αναφερθώ στα πολιτικά, αλλά οπωσδήποτε και η πολιτική κατάσταση ε, τα, τα μάλα επηρεάζει την ε, κατάσταση της ε, ασφαλείας. Το μήνυμα της Πρίστινα είναι ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα πρέπει να συμμετάχουν στο διάλογο. Πέστε τους κατηγορηματικά ότι αυτό είναι απαράδεκτο και το υπογραμμίζω το απαράδεκτο γιατί μετά η Σερβία θα πει εγώ θέλω και τη Ρωσία και μετά αντί για διάλογο τέτοιο θα ξεκινήσουμε ένα ε, ε, ε, διεθνή θα ξεκινήσουμε μια διεθνή διαδικασία ευρύτατη θα πρέπει να ενισχύσουμε τον ρόλο μας. Δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα από μόνοι τους αν δεν τους πρόξουμε, δεν τους πιέσουμε εμείς και το λέω αυτό γιατί δεν πιστεύω ότι εμείς τα κάνουμε, κάνουμε αρκετά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που μπορεί να χτυπήσει από την ευρωπαϊκή πλευρά το χέρι στο τραπέζι και να τους πει έτσι είναι και όχι αλλιώ. Νομίζω ότι τέτοιο ρόλο θα πρέπει να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στρατηγός ε, πολύ πιο προσγειωμένος ε, ήταν μιλώντας ε, για κάποιες δυνατότητες, κάποια ενδεχόμενα. Εάν ο στρατός του Κωσυφοπεδίου βρίσκεται στα βόρεια ας πούμε θα παρέμβει κάποια στιγμή. Ξέρετε ότι ο στρατός του Κωσυφοπεδίου θα τοποθετήσει οπωσδήποτε κάποια ε, τμήματα του στο βόρειο Κωσυφοπέδιο. Στρατηγέ, μπορείτε να μας πείτε τι δυνατότητες έχετε σε, αυτές, αυτήν την περίπτωση. Ξέρουμε ότι στο Βελιγράδι υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες είναι ήδη έτοιμες να ξεκινήσουν επιχειρήσεις στο Βόρειο στην Πρίστινα έχουν γίνει επεισόδια με τα οποία θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν ε, σε μέγιστο βαθμό επαγρύπνησης. Εντάξει, δεν θέλω να προκαλέσω πανικό, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να πάρουμε την κατάσταση πολύ πιο σοβαρά και να είμαστε πολύ πιο δραστήριοι και ε, να ανασκουμποθούμε και να κάνουμε κάτι. Ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Έντουαρτ. Είναι απόλυτα σαφές αυτό που λες. Είσαι σαφής και οι ερωτήσεις σου είναι σαφέστατες. Ο κύριος Σελίμωβιτς. Ευχαριστώ. Και ευχαριστούμε πολύ ε, για την ε, αξιολόγηση της κατάστασης. Ε, συμφωνώ με πολλά από αυτά που είπατε. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Όπως και ο κύριος Κούκαν, βλέπω ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική, όχι απαραίτητα με τα ίδια στοιχεία, αλλά γιατί έχουμε φτάσει πλέον σε μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, υπάρχει καχυποψία ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κωσυφοπαίδιο. Ε, υποσχεθήκατε την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Τώρα πιστεύω ότι θα πρέπει από τη στιγμή που και το Κοινοβούλιο μέσω της Επιτροπής του πήρε κάποιες αποφάσεις να πούμε και στην Κομισιόν να κάνει το ίδιο. Λένε λοιπόν αυτοί, ορίστε εμείς κάναμε ό,τι μας ζητήσατε αλλά δεν μας δώσατε αυτό που είχατε υποσχεθεί και τώρα δεν σας, ε, δεν σας ε, πιστεύουμε. Ε, ε, ναι, ε, και από την δική τους μεριά λένε εντάξει εμείς λέμε ότι θα μειώσουμε τους δασμούς μας, πιστεύετε. Άρα υπάρχει καχυποψία, έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ αυτών και ημών. Θα ήθελα να ενθαρρύνω πραγματικά το Συμβούλιο, με την ευκαιρία που έχω το λόγο, ε, να ακολουθήσει την αξιολόγηση του Κοινοβουλίου ε, και της Επιτροπής μας για τα θέματα ε, αυτά. Αυτά τα οποία ζητήσαμε, απαιτήσαμε από το Κωσυφοπαίδιο, τα παρέδωσε. Άρα και από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να παραδώσουμε. Εάν δεν θέλουμε να συνεχιστεί αυτό το ολιστηρό μονοπάτι της καχυποψίας η αξιολόγηση της κατάστασης όσον αφορά την ασφάλεια. Γίνονται συζητήσεις ε, για ανταλλαγές ε, εδαφών. Και αυτό ανακύπτει ξανά από την ε, Προεδρία και μερικές φορές και από εκπροσώπους του Υπουργείου Αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών. Ήμουν πέρσι εκεί, ξέρω τι συζητάει ο κόσμος και πρέπει να του φέρνουν ρίγη αυτές οι συζητήσεις. Στο κοσυφοπαίδιο λένε πάντα «Ναι, ναι, έχουμε συμφωνία, η κατάσταση είναι υποέλεγχο, αλλά εάν σκεφτεί κανείς τι θα μπορούσε να συμβεί αν κάτι τέτοιο προχωρήσει, τότε θα δημιουργηθεί πραγματικά μια κατάσταση ασφάλειας που θα είναι περίπου, περίπου στα όρια της ε, έκρηξης. Γιατί αυτά τα εδάφη δεν είναι ξεκάθαρα από εθνοτική πλευρά άποψη στο Κωσυφοπέδιο δεν είναι στο βόρειο τμήμα, δεν είναι μονάχα Σέρβοι ε, και από την άλλη πλευρά στην Κοιλάδα δεν είναι μονάχα ε, ε, εθνοτικά Αλβανοί. Δεν είναι ξεκάθαρη εθνοτικά η κατάσταση δηλαδή. Επομένως θα πρέπει να αξιολογήσετε πολύ σοβαρά τους ενδεχόμενους κινδύνους που θα επιφέρει η συνέχιση μιας τέτοιας κατάστασης. Εντάξει, η ιδέα του διαλόγου και των συζητήσεων είναι πολιτική. Δεν, λέω, δεν σας ρωτώ εάν σας αρέσει ή όχι. Ε, σας ρωτώ εάν βλέπετε ποιος μπορεί να είναι ο αντίκτυπος στην ασφάλεια αυτών των ε, ε, συνομιλιών. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Σελίμοβιτς. Έχω ακόμα δύο μιλητές. Παρακαλώ σύντομα όμως για να ακούσουμε και τις απαντήσεις. Θα μιλήσω ισπανικά. ο επόμενος ομιλητής. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Θέλω να ευχαριστήσω τους ομιλητές μας για τις πληροφορίες που μας έδωσαν για ένα θέμα που για τη χώρα μου είναι και αμφιλεγόμενο αλλά και σημαντικό γιατί είμαι Ισπανός Ευρωβουλευτής και είναι ένα μία από τις χώρες, η Ισπανία, που δεν αναγνωρίζει ως κυρίαρχο κράτος το Κωσυφοπαίδιο. Μας απασχολεί πάρα πολύ η κατάσταση και συμφωνώ με τους δύο προηγούμενους ομιλητές για την ανησυχία λόγω των αυξανόμενων εντάσεων. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε την οικονομική βιωσιμότητα ενός κράτους το οποίο είναι αδύναμο, που εξαρτάται από τους πιστωτές της Παγκόσμιας Τράπεζας για την ανοικοδόμηση και την ανάπτυξη και που έχει σοβαρά προβλήματα διαφθοράς, ε, δεν έχει διαφάνεια και που ε, επιδίνωσε την, τις εντάσεις που υπάρχουν με τη Σερβία λόγω των δασμών που αναφέραν διάφοροι ομιλητές. 100% αύξηση των δασμών στα σέρβικα προϊόντα. Επίσης, ε, η δήλωση του Δεκεμβρίου του 2018 για τη δημιουργία ενό στρατού μα ανησυχεί πάρα πολύ, δηλαδή ενό μια στρατιωτική δύναμης με 5.000 στρατιώτες, ε, το οποίο έρχεται σε αντίφαση με το ψήφισμα του ΟΗΕ 1244. Αυτές είναι οι βασικές ερωτήσει μου. Τι θέση έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην δημιουργία μια στρατιωτική δύναμη, ενό στρατού κοσοβάρικου. Επίσης, ε, χαιρετίζω ε, την ε, K4. Ε, επί 10 χρόνια 22.000 Ισπανοί στρατιώτες συμμετείχαν στην δύναμη αυτή. Μας ανησυχεί η ριοσπαστικοποίηση του πολιτικού Ισλάμ. Το 2017 διαβάσαμε μια έκθεση του προγράμματος του ΟΗΕ για την ανάπτυξη που μιλούσε για την φοβερή ανάπτυξη που έχουν τα ισλαμικά γκρουπ, οι ισλαμικές, ισλαμικές ακραίες ομάδες στο σκοσφοπέδιο. Αυξάνεται ο Ισλαμισμός, ο ακραίος Ισλαμισμός η ριζοσπαστικοποίηση κυρίως ε, ξεκινώντας από, τις, ε, από τα τζαμιά. Είδαμε επίσης ε, στην Επιτροπή για την Τρομοκρατία που δημιουργήσαμε στο Κοινοβούλιο ε, ότι συχνά η Σαουδική Αραβία ουσιαστικά υποβοηθάει την επέκταση αυτού του Ισλάμ έτσι πολύ ρηξικέλευτου χαρακτήρα θα πρέπει να μιλήσουμε τη Σαουδική Αραβία για να σταματήσει να το κάνει. Λοιπόν, Υπάρχει συνειδητοποίηση αυτού του κινδύνου για την επιστροφή δεκάδων ε, Αλβανών και Κωσοβάρων που ήταν στη Συρία και πολέμησαν εκεί με τις διάφορες δυνάμεις και μπορεί να επιστρέψουν στην Ευρώπη. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό, ο κύριος Σόλτες. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ συγγνώμη, καθυστέρησα πολύ. Ήμουνα πρόεδρος της ε, ομάδας των σκιωδών εισηγητών και δεν μπορούσα να έρθω πριν. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κούκαν και τον κύριο Σελίμοβιτς. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το, την κατάσταση ασφάλειας στο κοσμοπέδιο για διάφορους λόγους και ο ένας από αυτούς δεν αφορά το ίδιο το κοσμοπέδιο, ο ένας από αυτούς. Θα ήθελα επίσης να τονίσω το θέμα της απελευθέρωσης του καθεστώτος θεωρήσεων. Υποσχεθήκαμε πολλά στους Κωσοβάρους και δεν διακρίνουν οι Κωσοβάροι έτσι, στο δημόσιο βίο τους ανάμεσα στο Κοινοβούλιο, την Κομισιόν, το Συμβούλιο κτλ. Ένα ε, είμαστε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Και με αυτή την προσέγγιση φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να είμαστε πρόσδεκτοι πια στο κοσφοπέδιο. Αν δεν αλλάξουμε τη στάση μας και δεν του στείλουμε ένα σαφές μήνυμα, ε, κάνουμε διάκριση εμείς απέναντι στην Σερβία και στο Κοσφοπέδιο. Γιατί οι Κοσοβάροι έχουν την αίσθηση ότι αντιμετωπίζουμε διαφορετικά τη Σερβία από το Κοσφοπέδιο. Και τους έχουμε κάπου εκεί στην ερημιά μόνους τους, στο απότατο μέλλον κτλ. Δεν εκπλήσωμε λοιπόν που αντιδρούν έτσι. με αυτές τις αντιδράσεις που δεν είχαν ξανασυμβεί. Ε, και συμπεριλαμβανομένου εδώ και των φόρων που έπληξαν κυρίως στη Βοσνία. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι διπλωματικά μέσα έχουμε για να τους πείσουμε να πείσουμε το Συμβούλιο να δώσει το πράσινο φως ή τουλάχιστον να τους δώσει ένα μήνυμα ότι η απελευθέρωση το, από την υποχρέωση θεωρήσεων δεν είναι όνειρο, αλλά είναι πραγματικότητα, γιατί το χρειαζόμαστε αυτό για τη σταθερότητα στην περιοχή. Με ανοιχτό διάλογο θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση και να μειωθούν αυτές οι εντάσεις που δεν μπορείτε απλώς να τις ε, αισθανθείτε, ε, να τις ψυχανεμιστείτε, αλλά να τις ε, δείτε κιόλας. Και συμφωνώ με αυτά που είπε με, υπό την επίσημη ιδιότητά του ο υποστράτηγος για το κοσφοπέδιο. Αν αυτή η παγωμένη ένταση ε, παραμείνει ως τέτοια για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πού μπορεί να οδηγήσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ στο τέλος ε, να αναφερθώ σε ένα σχολείο του υποστρατηγού Νταντάριο ότι ακόμα και η εντύπωση μιας ε, ρήξης ανάμεσα στο Κωσοφοπέδιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι επικίνδυνη υπό αυτές τις ε, συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα κάποιο σχόλιο από τον κύριο Κάλαν. Τι γίνεται εάν ας πούμε αυτήν την εβδομάδα στο πλαίσιο της ε, συνάντησης στο ΝΑΤΟ συζητηθεί ε, το τι μπορεί να γίνει για να αποφύγουμε αυτόν τον κίνδυνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ενημερώσω ότι η διερμηνία θα έχουμε μέχρι τις 12.30, οπότε δεν έχετε πολύ χρόνο να απαντήσετε. Μπορούμε μετά να συνεχίσουμε, αλλά χωρίς διερμηνία. και μπορείτε να απαντήσετε με τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις ή όπως θέλετε, όπως πριν. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Να πω καταρχά ευθύ εξ αρχή πω ευχαριστώ το Κοινοβούλιο για τη στήριξή του, διότι μα έχει βοηθήσει πάρα πολύ η βοήθεια αυτή και ελπίζουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε τις ε, στήριξή σα και στο μέλλον. Τώρα, ε, να πάρω τι ερωτήσει από την αρχή. Αναφερθήκατε πολύ στους δασμούς και γιατί δεν δεν καταλαβαίνουν το μήνυμα. Γιατί, και, γιατί το μέτρο αυτό χρειάζεται σαφήνεια. Να σας ε, πω πως ε, είναι ένα μέτρο που κατάφερε να ενώσει ε, τον κόσμο μέσα σε μια πολύ τεταμένη πολιτική ατμόσφαιρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μέχρι και πολιτικοί που στην αρχή ήταν αρκετά επιφυλακτικοί για τους δασμούς έπρεπε να συμφωνήσουν με ένα αρκετά δημοφιλές μέτρο το οποίο θεωρούν ένα μέτρο ε, που είναι η μόνη λύση για να αντιμετωπίσουν μία προκλητική, επιθετική συμπεριφορά της Σερβίας. Και αυτό τους έδωσε αυτοπεποίθηση. Και δεν νομίζω ότι η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ε, ήταν αρκετά έντονη στην ε, διατύπωσή τη, αλλά και εκείνη και ο Πίτροπος Χάν μέσω επιστολών έχουν καταστήσει σαφή την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωση για τα μέτρα αυτά. Παρά το γεγονός ε, λοιπόν ότι το μήνυμα αργεί να φτάσει, νομίζω ότι τελικά έχει ακουστεί από τους ε, εταίρους μας στην Πρίστινα. Και υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι το μήνυμα αυτό ε, ίσως τους κάνει να ξανασκεφτούν τα μέτρα αυτά. Ίσως δούμε κάποια αλλαγή στο πρόσεχες μέλλον. Αλλά όπως είπα και πριν, συνεργαζόμαστε με τους εταίρους μας και έχουμε ευθυγραμμίσει την στάση μας σε όλα τα επίπεδα. Είμαστε κατά των μέτρων αυτών λοιπόν και θέλω να πιστεύω πως ε, στο τέλος θα μας ακούσουν. Ε, σίγουρα δεν ε, μας υποτιμούν, διότι η στάση μας ήταν έντονη και σκληρή. Και να σας πω επίσης πως για το κοσυφοπαίδιο αυτό το πρόγραμμα του στρατού είναι κάτι που τους ενώνει, είναι κάτι που έχει μεγάλη απήχηση στο λαό και σίγουρα δεν είμαστε ευχαριστημένοι, το έχουμε καταστήσει και αυτό σαφές και θα φροντίσουμε να γίνει ακόμα πιο ορατό. Και εδώ επίσης συμφωνούμε απόλυτα με το ΝΑΤΟ, είμαστε ευθυγραμμισμένοι και θα συνεχίσουμε την συνεργασία και εδώ στις Βρυξέλλες και σε επίπεδο Γενικού Γραμματέα και Ήπρα της Εκπροσώπου, αλλά και επιτόπου. Η ΚΕΙΦΟΡ δηλαδή θα είναι η φωνή μας στο κοσφοπέδιο. Τώρα η απελε... σχετικά με την απελευθέρωση. Συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλιά σας. Κατανοώ βέβαια την αγανάκτηση ε, στο κοσυφοπαίδιο σχετικά με την απαλλαγή αποθεώρηση, αλλά πρέ... χρειάζεται πολλή δουλειά ακόμα. Έχουν όντως ε, τηρήσει τις ε, δεσμεύσεις τους, όμως υπολείπονται πολλά ακόμα και πρέπει να συνεχίσουν να καταπολεμούν το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και ε, το κράτος δικαίου έχει ακόμα, είναι ένα, ε, ένας τομέας στον οποίο έχουν ακόμα χαμηλές επιδόσεις. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουν οι προσπάθειες και μόλις ε, είναι έτοιμοι θα τους χορηγηθεί και η απαλλαγή από την έκδοση θεώρησης. Σε ό,τι αφορά το διάλογο και τις Ηνωμένε Πολιτείε, πράγματι έχουν γίνει αυτές οι δηλώσεις από την Πρίστινα, τους κατηγόρησαν ε, ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν καταλάβει σχεδόν ε, τη χώρα και τις προσπάθειες, όμως υπάρχει ένας διάλογος, θέλουμε να συνεχιστεί Δεν νομίζω πως παραμεριζόμαστε καθόλου και η είπατε εκπρόσωπος ε, έχει εργαστεί πάρα πολύ για να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος και έτσι κι αλλιώς η πλευρά των ΗΠΑ ε, ήταν ε, ανοιχτή και σε επικοινωνία μαζί μας. Μπορώ να σταματήσω όμως εδώ και να δώσω το λόγο στον David για παραπάνω πληροφορίες. No,